σε 9 το πρωί, το απόγευμα και το βράδυ. Η μερική διάταξη έχει δημοσιευθεί στο ανάλογο εγγράφο και στο ίντερνετ. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Καληνύχτα.